Λοιπόν, λέει ο πρόεδρο. Με 20 λεπτά καθυστέρηση θα πάμε στο σημείο 6, πολύ σύντομα όμως, όπως είχαμε συμφωνήσει. Σύντομη ενημέρωση σχετικά με την αντιπροσωπεία μας ε, στην Ουάσιγκτον, 17 συναδελφοί ΑΦΕΤ, ΣΕΝΤΕ και στη Γενική Συνέλευση 23 με 27 Οκτωβρίου 27 και 31 μάλλον Οκτωβρίου και με τους τις προέδρους της ε, ΑΦΕΤ, ΣΕΝΤΕ Κεντροά Ήταν η πρώτη επίσημη αντιπροσωπεία της δικής μας Επιτροπής ε, στην Ουάσιγκτον και αυτό δείχνει το, τη σημασία που δίδουμε στην διατλαντική συνεργασία και σχέση στη Νέα Υόρκη. Είχαμε συνομιλίες και με τον κύριο Γκουτέρες και σε επίπεδο πρέσβεων. Στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών συναντήσαμε την Ινδική μόνιμη αντιπροσωπεία, το οποίο έδωσε και διαβίβασε το μήνυμα ότι έχουμε στόχους ενισχυμένης συνεργασίας και συνομιλίας για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το Συμβουλίο Ασφαλείας, το σύστημα της πολυμέρειας επί τη βάση κανόνων και διατάξεων, την επίτευξη συνένευσης ε, στην διεθνή κοινότητα και την αποφυγή αποκλήσεων και κατακαιρματισμού, να παραμείνουμε δηλαδή μια συνεκτική ομάδα στο, στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με μια σαφέστατη τοποθέτηση πολιτικής εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καλήσαμε, και, καλέσαμε μάλλον και τους, τις αντιπροσωπείες μας στα Ηνωμένα Έθνη, όποτε επισκέπτονται τις Βρυξέλλες να επισκέπτονται και μας, να μας ενημερώνουν τις, τις σχεδιαζόμενες με συγχωρείτε δραστηριοτήτες για, την... για τον εορτασμό της ε, επαιτίου των Ηνωμένων Εθνών του χρόνου στην Ουάσιγκτον συναντήσαμε πέντε μέλη της Γερουσίας παρά τις διαδικασίες impeachment που δημιούργησε κάποια προβλήματα χρονοδιαγράμματος. Επίσης μέλη του Κοινοβουλίου, του Κογκρέσου. Συζητήσαμε για τη Βενεζουέλα με τον κύριο Έλιοτ Άμπραμς, ειδικά απεσταλμένο και υπεύθυνο για τα θέματα Τη προσέγγιση για τη Βενεζουέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών είδαμε ότι η συνεργασία με τους Αμερικανούς είναι δυνατή παρά τις δυσκολίες της τελευταίας ε, στα θέματα ιδιαίτερα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημο... αρχών της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά στην Κίνα, όλοι σημειώσαμε την απόφαση της απονομής του βραβείου Σαχάροφ στον, στον Τότι. Επίσης ε, σημειώθηκαν τα θέματα των Δυτικών Βαλκανίων. Εμείς πάντως δηλώσαμε την ε, θετική μας τάση για τα θέματα διατλαντικής ε, συνεργασίας Επίσης συναντηθήκαμε με το National Endowment for Democracy. Όλες αυτές ήταν πολύ θετικές συνομιλίες με τροφή για σκέψη για το μέλλον των ε, διατλαντικών μας ε, σχέσεων. Αυτά εν συντομία να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που συμμετείχαν στην επίσκεψη, στην αποστολή και να, προσέψω, να προσθέσω απλώς προσωπικά ότι καμιά φορά μας εκπλήσει ε, πώς μας μεταχειρίζονται ως μέλη του Κοινοβουλίου όταν προσπαθούμε να εισέλθουμε σε κυβερνητικά κτίρια. Νομίζω ότι αν μεταχειριζόμασταν έτσι, αν συμπεριφερόμασταν έτσι σε μέλη της γερουσίας των ΗΠΑ, αυτό θα, είχε, θα δημιουργούσε σκιές στη σχέση μας. Βεβαίως προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πέντε λεπτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σιμοτσέβιτς, θέλετε κάτι να πείτε. Ε, δύο λόγια απλώς, Πρόεδρε. Όλοι οι θεσμικοί φορείς ε, που επισκεφθήκαμε ε, μάλλον υπήρχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με, το, με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ ιδιαίτερα στα θέματα των επιθέσεων ε, στον κυβερνοχώρο, γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα, λέει ο μιλητή. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Αν δεν έχουμε άλλο σχόλιο μπορούμε να πάμε στο σημείο